Ωραία, όπως βλέπω έχουν φτάσει μερικοί συνάδελφοι εκτός από όλους τους συνεργάτες μας στην Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε Μπορούμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση της μελέτης σε σχέση με την πρόθεση της καινοτομία στο διαδίκτυο και το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτική ζωή. Όσον αφορά το θέμα αυτό, θα μιλήσουν σήμερα ο Τζόναθαν Κέιφ και ο Μάρκ Βαν Λίσχαουτ. για 15 λεπτά ο καθένας. Μετά θα έχουμε 20 λεπτά περίπου για ερώτα απαντήσεις και μετά 5 λεπτά για τις απαντήσεις. 11, 12, 15 το πολύ. Το 15 λεπτά που σας είπα είναι τα πολλά. Μπορείτε να μιλήσετε και λιγότερο αν θέλετε. Αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο. Θα ξεκινήσει ο κύριος ε, Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μάρκ Φαν ε, Είμαι από την Ολλανδία. Ε, θα Έχω ετοιμάσει όμως την παρουσίαση στα αγγλικά. Ε, θα την παρουσιάσω λοιπόν στα αγγλικά. Είμαι ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης που βρίσκεται μπροστά σας. Σύντομα θα σας παρουσιάσω μια σειρά διαφανειών και θα επικεντρωθώ στα συμπεράσματα. Είμαι αρκετά βέβαιος ότι έχουμε κάνει ε, όσα μας ζήτησε το ε, Κοινοβούλιο όσον αφορά τη μεθοδολογία, αλλά θα επικεντρωθώ στο τμήμα μεθοδολογίας. Ορίστε οι ερωτήσεις που μας ε, έθεσε το Κοινοβούλιο. Να συνοψίσουμε τις εγγύησει για την ιδιωτική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι τάσεις και εντάσεις και ποιες είναι οι δυνατότητες να προωθήσουμε την ε, καινοτομία και ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο διαδίκτυο, ε, ε, σεβόμενοι όμως τον, την ιδιωτική ζωή. Κάναμε το εξή. Είπαμε ότι αν κοιτάει κανεί την καινοτομία στο διαδίκτυο και την ιδιωτική ζωή, θα πρέπει να κοιτάξει κανεί την σχέση εδώ. Θα πρέπει να δούμε πώ προωθείται η καινοτομία από την ιδιωτική ζωή. Θα πρέπει να δούμε πώς εμποδίζεται η καινοτομία από το δικαίωμα στην ε, ιδιωτική ζωή και αντίστροφα θα πρέπει να δούμε πώς ε, προωθείται η ιδιωτική ζωή, ο ιδιωτικός βίος από την καινοτομία και πώς ε, εμποδίζεται από την καινοτομία. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία τετραπλή μια τετραπλή σχέση. Στην έκθεση θα βρείτε λεπτομέρειες της προσέγγισής μας. Εξετάσαμε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, οι οποίες ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Κοιτάξαμε την διαφήμιση στο διαδίκτυο, το υπολογιστικό νέφος RFID, και μία πέμπτη περίπτωση εξετάσαμε. Είχαμε ένα εργαστήριο πυροχνωμόνων στο οποίο καλέσαμε ε, ανθρώπους από αυτούς τους διάφορους τομείς ε, και τους ζητήσαμε να μας, ε, πούν, να μας περιγράψουν τη σχέση αυτή ανάμεσα στην κερατομία και το ιδιωτικό απόρριτο και τελικά παρουσιάσαμε την έκθεση που έχετε μπροστά σας. Όσον αφορά το νομοθετικό τοπίο, ε, δεν ε, χρειάζεται να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στον τομέα αυτών. Ε, βασικά, η οδηγία περί ιδιωτικού βίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βασική εδώ. Υπάρχουν όμως και άλλες οδηγίες που μας ενδιαφέρουν. Ε, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι ο, κανονισμός, ο προτινόμενος ε, κανονισμός του Συμβουλίου ε, που σκιαγραφεί τι μπορεί να αναμένεται από τις επιχειρήσεις όσον αφορά το διαδίκτυο και το ιδιωτικό απόρριτο. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε μια σειρά θεμάτων, να δούμε πώς μια πώς οι οδηγίες αυτές επηρεάζουν ε, την ε, καινοτομία και, την, ε, και τον ιδιωτικό βίο ανθρώπων. Ένα από τα μία από τις, ε, ε, ένα, ένα από τα γεγονότα ε, των... Υπάρχουν πολλά γεγονότα μάλλον των τελευταίων ετών που σας παρουσιάζουν πόσο πολύπλοκη είναι η σχέση αυτή. Αρκεί να σας, αναφερθώ, αρκεί να σας αναφέρω κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, την Google. Υπάρχει το Google Street View και αρκετές χώρες απαγόρευσαν την υπηρεσία Street View, κάτι που οδήγησε και σε κατάρρευση των των εξυπηρετητών στην ε, Γερμανία, των σερβερ στη Γερμανία. Ε, εάν εξετάζουμε την καινοτομία θα πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο ε, την τεχνολογική αλλά και την θεσμική καινοτομία. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό ε, παράγοντα στο ιδιωτικό απόρριτο και στο πώς πραγματοποιείται η καινοτομία. Θα πρέπει να δούμε πώς οι χρήστε παίζουν ρόλο εδώ. Ιδιαίτερα διότι αν κοιτάξουμε τα κοινωνικά μέσα όπως το Facebook ε, θα δείτε ότι ο χρήστης ε, ε, παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και το πώς λαμβάνουν υπόψη το ιδιωτικό απόρριτο. Αυτή λοιπόν ήταν η προσέγγιση μας. Είναι αρκετά πολύπλοκη η προσέγγιση μας. Προσπαθούμε στην έκθεσή μας να δείξουμε ότι όλα τα στοιχεία αυτά, αν τα δούμε συνδυασμένα διαφωτίζουν τη σχέση ανάμεσα στην καινοτομία και το ιδιωτικό απόρριτο και το πώς αναπτύσσεται η σχέση αυτή. Στην έκθεσή μας, ε, λοιπόν, προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε πώς ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις πτυχές αυτές. Ε, δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε από το συμπέρασμα ότι το ιδιωτικό απόρριτο απειλείται από την καινοτομία. Ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στην καινοτομία και το ιδιωτικό απόρριτο και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε αυτό ε, με μια σειρά υποσυμπερασμάτων. Ε, γενικά, αν δούμε ε, ποιοι βρίσκονται ε, στην αιχμή νέων ε, υπηρεσιών, βλέπουμε ότι οι πολλά δεδομένα είναι ταυτοποιήσιμα. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επίσης είπαν ότι τα ε, προσωπικά δεδομένα είναι το πετρέλαιο της ε, νέας ε, παγκόσμιας οικονομίας. Όλες αυτές οι υπηρεσίες κάνουν χρήση των προσωπικών δεδομένων ώστε οι υπηρεσίες να είναι, όσο, είναι προσαρμοσμένες στο άτομο βρήκαμε πολλά παραδείγματα του πώς η καινοτομία μπορεί να προωθήσει το ιδιωτικό απόρριτο και τις σχετικές τεχνολογίες, αλλά θα το αναπτύξουμε και αυτό. Και όσον αφορά τη τεχνολογία και τις επιχειρηματικέ πρακτικές και όσον αφορά τις εμπειρίες μας παντού, υπάρχουν κάποια παραδείγματα του πώς οι υπηρεσίες προσπαθούν να αναπτυχθούν Λαμβάνοντα υπόψη χαρακτηριστικά τα οποία ε, αυξάνουν το ιδιωτικό απόρριπτο, προστατεύουν το ιδιωτικό ε, και η τεχνολογία για την προστασία του ιδιωτικού απορρίτου μπορεί να αποτελούν παραδείγματα καινοτομίας, αλλά όλα αυτά δεν αντισταθμίζουν ε, ε, την αντίστροφη σχέση. Ε, επίσης, οι καινοτόμοι θεωρούν ότι το ιδιωτικό απόρριτο είναι ε, παράγοντας κόστους, ε, δεν το βλέπουν ως κάτι θετικό. Εάν συμπεριλάβουν το ιδιωτικό απόρριτο στα επιχειρηματικά μοντέλα τους, αυτό στοιχίζει. Αυτό ισχύει και όσον αφορά την τεχνολογία, αλλά και όσον αφορά την οργάνωση. Θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρίτου. Αυτό είναι θέμα οργάνωσης και στοιχίζει. Ε, κατόπιν έχουμε τα συμπεράσματα για τις ε, αναδυόμενες τεχνολογίες. Ε, κοιτάμε διάφορα παραδείγματα του πώς αναπτύσσονται οι τεχνολογίες αυτές, τι μας λένε για την τεχνολογία. Μας δείχνουν ότι η σύγκληση τεχνολογιών του διαδικτύου και άλλων και άλλες ε, αυξάνουν τα ε, προβλήματα ιδιωτικού απορρίτου. Ε, επηρεάζονται όλο και περισσότερο στις ομάδες. Αν κοιτάξουμε το υπολογιστικό νέφος ή τις υπηρεσίες που βασίζονται στον τόπο που βρίσκεται το πρόσωπο, οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται ταυτοποιήσιμα στοιχεία για να λειτουργήσουν. Έτσι, λοιπόν, οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τέτοιες λύσεις. έχουμε τα, γενετικά, τα γενικά δεδομένα και τα πιο προσωπικά. Ε, αν κοιτάξουμε τις ε, τεχνολογίες που είναι φιλικές ε, προς, που προστατεύουν το ιδιωτικό απόρριτο. Υπάρχουν εδώ κάποιες. Έχουμε κάποια παραδείγματα όπου η τεχνολογία και η προστασία του ιδιωτικού απορρίτου πάνε χέρι-χέρι. Γενικά όμως όλοι γνωρίζουμε ε, ότι υπάρχουν κάποια παραδείγματα ε, και στα κοινωνικά μίδια ε, όπου προβλέπεται η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι υπηρεσίε αυτέ ότι είναι δύσκολο ε, να γίνουν αποδεκτέ από ε, τις επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Ε, Όσον αφορά τις επιχειρηματικέ πρακτικές, ε, οι νέε επιχειρηματικέ πρακτικές ε, γενικά τονίζουν ε, την κερδοφόρα χρήση των προσωπικών δεδομένων άλλων και είναι ουσιαστικά το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης αυτής ότι τα, τα στοιχεία, εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να διέπεται η χρήση αυτή από κανόνες. Είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει κανείς ε, αποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα. Ε, έχουμε και πάλι την πίσω πλευρά του νομίσματος. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που προσπαθούν ε, να λάβουν υπόψη τους ε, τα στοιχεία αυτά, αλλά οι ε, καταναλωτές ε, δεν φέρονται πολύ διατεθειμένοι να πληρώσουν για κάτι τέτοιο. Την έκθεσή μας μπορείτε να τη διαβάσετε. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι αν κοιτάξετε τα πειράματα που πραγματοποιούνται στον τομέα αυτό όσον αφορά την επιχειριστική οικονομία, ο κόσμος μπορεί να προτιμάει μια υπηρεσία, αλλά μόνο εφόσον δεν στοιχίζει. Εφόσον στοιχίζει μια υπηρεσία, φαίνονται να μην προτιμάει προτιμούν οι καταναλωτές ε, την ε, υπηρεσία που προστατεύει καλύτερα το ιδιωτικό του απόρριτο. Έτσι, λοιπόν, αν κοιτάξετε τις, ε, τις έρευνες, ο κόσμος λέει ότι απαντάει ότι τον ενδιαφέρει το ιδιωτικό απόρριτο του. Αν δείτε τη συμπεριφορά του κόσμου όμως, θα διαπιστώσετε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ πολύ συγκεκριμένα, εάν έχουν επιλογή, θα επιλέξουν την επιλογή που προστατεύει το ιδιωτικό τους απόρριτο. Αυτό έχει την συνέπεια για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών ότι ε, μπορούν να αναπτύξουν υπηρεσίες ε, ε, που να προστατεύουν το ιδιωτικό απόρριτο. Στο συμπέρασμα 9 βλέπετε ότι οι κανόνες για την προστασία του ιδιωτικού απορρίτου παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά ε, αυτή τη στιγμή η, πιθανότητα να ε, εντοπιστεί κανείς ε, όταν ε, παραβιάζει την ε, προστασία του ιδιωτικού απορρίτου δεν είναι πολύ μεγάλη. Εάν είναι να υπάρξουν κάποια προστατευτικά μέτρα, ε, ουσιαστικά χρειάζεται κάποια παρέμβαση. Υπάρχει σαφής ανάγκη ε, και μάλιστα η ε, προστασία του ιδιωτικού απορρίτου συνήθως δεν αποτελεί αντικείμενο αυτό ελέγχου από τις επιχειρήσεις Αυτό ήταν ε, το δικό μου ε, κομμάτι της ε, παρουσίαση. 13 λεπτά μίλησα. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι τήρησα το χρόνο μου. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για τις συστάσεις προς το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Μάρκα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε να ακούσετε την παρουσίασή μας. Όταν μιλάω για συστάσεις στην έκθεση, κάναμε προσπάθειες ε, οι συστάσεις να εστιαστούν, να είναι εστιασμένες και να μπορούν να είναι εφαρμόσιμες. Συνεπώς δεν έχουμε μπει σε τεράστιο βαθμό λεπτομάρειες. Θα προσπαθήσω να ε, επικεντρω... να προκαλέσω κάποια συζήτηση, να δώσω κάποιο περιθώριο για συζήτηση. Η πρώτη σύσταση είναι ότι το ιδιωτικό ε, απόρριτο ω δικαίωμα προστατεύεται στον ευρωπαϊκό χώρο ω θεμελιώδη δικαίωμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, δεν μπορεί να καταργηθεί και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευση μέσω μηχανισμών τη αγορά. Από την άλλη, στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και σε ορισμένα μέρη τη Ευρώπη, μάλιστα, το ιδιωτικό απόρριτο είναι ένα οικονομικό δικαίωμα ή μάλλον οι ιδιωτικέ πληροφορίε έχουν οικονομική αξία. Και ένα από τα πράγματα που καθίσταται προφανέ είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση καθεστώτων. Στο ένα μέρο του κόσμου θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα και στο άλλο θεωρείται οικονομικό δικαίωμα. Και έτσι καταλήγουμε ενδεχομένω σε, μια κατάσταση όπου κανένα από τα δύο δικαιώματα δεν είναι προστατευμένο. Μπορούν να, να αποτελέσουν οι πληροφορίε αντικείμενο εκμετάλλευση βάσει οικονομικών συμφερόντων για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, το οποίο γίνεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο Μάρκ αναφέρει τον Google, δεν είναι μόνο το Streetfield και δεν είναι μόνο το κατά πόσο οι... μπορούν να δουν οι ληστές στο δικό σας ε, σπίτι, είδαμε και το G-Stumbler, ενώ παίρνουν φωτογραφίες κοιτούν μέσα από μία ασφαλή ασύρματα δίκτυα, λαμβάνουν όλε τι πληροφορίε και τα ανεβάζουν σε σερβέρ στι ΗΠΑ. Εδώ και πολλούς μήνες ανακαλύψαμε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και ότι αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το ιδιωτικό απόρριτο είναι ατομικό δικαίωμα, αλλά δεν είναι πραγματικά ατομικό δικαίωμα. Όταν χρησιμοποιώ υπολογιστικό νεφο, οι δραστηριότητε του παρόχου τη υπηρεσία νεφου είναι πληροφορίε σε σχέση με το τι κάνω εγώ. Είναι δηλαδή προσωπικέ πληροφορίε για μένα, αλλά είναι ε, νόμε πληροφορίε αυτού του ατόμου. Ε, αν εμεί οι δύο συζητάμε κάτι, είναι από κοινού ιδιωτικέ αυτέ οι πληροφορίε. Εγώ έχω ένα νομικό, νόμιμο συμφέρον το να μην ε, θέλω να μάθει κάποιο ότι μιλάω με εσά και εσεί επίση μπορεί να μην θέλετε να μάθει κάποιο ότι μιλάτε με μένα. Ποιο θα προστατεύσει τι πληροφορίε, ποιανού είναι αυτέ τι πληροφορίε ε, ενό από εμά. Αν εγώ δεν συλλέξω πληροφορίε που σα εντοπίζει, αναγνωρίζει ω άτομα, αλλά σα αναγνωρίζει μεταξύ ενό συγκεκριμένου πλήθου ατόμων. Για παράδειγμα, ο ταχυδρομικό μα ο ταχυδρομικός σα κώδικα, τα εθνικά σα χαρακτηριστικά, τα δημογραφικά σα μοτίβα, όλα αυτά μπορούν να καταλήξουν σε πράγματα ανησυχητικά. Σε περίπτωση που μπορέσω να σας αναγνωρίσω, μπορώ να αποκτήσω τα περισσότερα σας στοιχεία, ε, μπορεί να περιορίσω την ελευθερία δράση σας και ούτω καθεξής. Ενώ λοιπόν στην αρχή το θεωρώ ότι είναι ατομικό αγαθό. Έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι το δυτικό απορρίτο αφορά μόνο την προστασία των δεδομένων. Αυτό προέρχεται από παλιότερε τεχνολογίε όπου πολλά πράγματα γίνονταν εκτό σύνδεση offline, όπου το ιδιωτικό απορρίτο είχε σχέση με την ταυτότητά μου. Η ταυτότητά μου ήταν μια σειρά από αρχεία, μητρώα. Αλλά όταν είμαστε online, οι πληροφορίε που δημιουργούνται, μόνο από το γεγονός ότι εγώ μπαίνω στο διαδίκτυο. Ε, δηλαδή αν έχω μια ιστοσελίδα, όταν μπαίνω σε μια ιστοσελίδα μου ζητούν κάποιες πληροφορίες. Ανάλογα με τις πληροφορίες που δίδω εξαρτάται η επόμενη οθόνη που θα δω και οι συνέπειες είναι ότι η ελευθερία δράσης μου και το ιδιωτικό χαρακτηριστικό των δράσεών μου περιορίζεται από το ίδιο το σύστημα. Μπορεί λοιπόν να μην έχει να κάνει με δεδομένα, αλλά με άλλα στοιχεία, όπως το παλιότερο δικαίωμα ιδιωτικού απορρίτου, το δικαίωμα του να με αφήσουν ήσυχο, το να μην έχω την αίσθηση ότι με παρακολουθούν διαρκώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συστάσεις που θα πρέπει ίσως να λάβουμε υπόψη κατά πόσο δηλαδή τα αριθμιστικά και νομοθετικά μας πλαίσια είναι ο τρόπος ε, ε, ε, ε, λαμβάνω όλα αυτά υπόψη με τον κατάλληλο τρόπο. Ένα άλλο πράγμα, όπως είδαμε με τους νόμους για τα cookies, ε, η ενημερωμένη συνένεση είναι ένα ε, σωστός τρόπος για να βασίσουμε την όλη διαδικασία. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι κάνουν ενημερωμένε επιλογέ για το τι πράττουν, τότε ό,τι επιλέξουν να πράξουν είναι εντάξει. Και από τη δουλειά του κράτου να διασφαλίσει ότι κατανοούν αυτό που κάνουν. Αλλά στις πληροφορίες των πληροφοριών που ρέουν μέσω του διαδικτύου και που μπορεί να επιβιώνουν όχι στις αρχικές τους ε, μορφές αλλά υπό τη μορφή επικρίσεων κατά εμάς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε νέες, οι κρίσεων για το άτομό μας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε νέες τεχνολογίες που δεν είχαν καν επινοηθεί τη στιγμή καταγραφής των πληροφοριών. Διότι το διαδίκτυο έχει τεράστια άπειρη μνήμη για άπειρο χρονικό διάστημα. Μπορεί λοιπόν να, ε, να μην γνωρίζουμε σε τι συνονούμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα στις ζωές τους. Το ιδιωτικό μου απόρριτο ως ενήλικα ε, παραβιάστηκε όταν εγώ ήμουν ένας νέος, ε, μπορεί να παραβιαστεί όταν εγώ, επειδή εγώ ήμουν ένας νέος ακτιβιστής. Ε, μπορούμε να περάσουμε κανόνες για το δικαίωμα του να ξεχαστούμε, αλλά εάν δεν τεθούν σε εφαρμογή οι άνθρωποι ε, κάνουν ενημερωμένε επιλογέ, αλλά μπορεί να μην ξέρουν ακριβώ τι επιλογή κάνουν. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όταν επιβάλλουμε τέτοια πράγματα όπω την ενημερωμένη συνένεση δημιουργούνται φραγμοί εκτό από ε, δικαιώματα και ευθύνε. και πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αναλογική, αποτελεσματική και σωστά καταμερισμένη. Σήμερα το πρωί αποφασίστηκε από το ICL στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι η υλοποίηση τη οδηγία για τα cookies δεν σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεις τη συνένεση κάθε συμβαλόμενου μέρους με κάθε ιστοσελίδα που έχει cookies, αλλά μόνο σε σχέση με κάποιες πληροφορίες που θεωρούνται εκ των προτέρων ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτό αλλάζει τον τρόπο υλοποίησης του νόμου και δεν είναι ομοιόμορφη αυτή στον ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και οι πτυχές της ενιαίας αγοράς, διάφορες άλλες πτυχές που αφορούν την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαι ακόμη στο πρώτο σημείο, αλλά σύντομα θα το ολοκληρώσω. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η λύση μπορεί να μην είναι η ψήφιση νόμων, αλλά το να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα έχουν εργαλεία που του προσφέρουν έλεγχο των πληροφοριών του. Υπάρχει τώρα μια διαφορά μεταξύ των εργαλείων που λαμβάνουν τα άτομα, οι πολιτικέ ιδιωτικού απορρίτου, των Google, του Facebook, μεγάλων εταιριών και τη ικανότητα των ανθρώπων να κατανοήσουν αυτά τα εργαλεία και να τα εφαρμόσουν. Από την άλλη έχουμε τεχνολογικές λύσεις όπως το Privacy by Design που εξορισμού δεν έχει επαρκή διαφάνεια και παρέχεται με διαφορετικούς τρόπους από τον κάθε πάροχο. Θέλουμε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στα νέα πράγματα που εμφανίζονται. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν ε, προκαταβάλουμε τα μοντέλα μας της ενημερωμένης επιλογής ε, τότε οι άνθρωποι ε, φοβούνται ή αντιδρούν υπερβολικά και μπορεί να χρειάζονται νομική προστασία. Τα εύλογα λοιπόν ε, μοντέλα, τα μοντέλα εύλογης απόφασης μπορεί να μην είναι το καλύτερος τρόπος. Το δεύτερο σύνολο συστάσεων μας έχει να κάνει με συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Θέλω απλά να σημειώσω για αυτό το θέμα ότι οι κανόνες που ψηφίζει οποιοδήποτε αρμόδιος φορέας δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν, εμπλέκονται και άλλα μέρη, τα ρυθμιστικές αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές, αυτορυθμιστικές αρχές, δημόσιες, την αλληλεπίδραση δημοσίων και ιδιωτικών αρχών. Υπάρχει το Harbor Provision. Ε, αυτό που συμβαίνει με αυτό είναι ότι το Υπουργείο Εμπορίου ε, προσυπογράφει την συμπεριφορά των παρόχων ίντερνετ, δηλαδή διερευνά παράπονα από ένα μέλος αυτού του οργανισμού κατά ενός άλλου μέλους της βιομηχανίας. Δεν παρακολουθεί και δεν επιβάλλει καμία νομοθεσία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Άλλοι τομεί όπου αυτό συμβαίνει είναι τομεί διένεξη πολιτικών, όπως περιβαλλοντική πολιτική. Ένας από τους τομεί που έχει θέματα απορρίτου στο διαδίκτυο είναι τα smart grid και οι έξυπνοι μετρητέ. Διότι λένε, μας λένε ποιο βρίσκεται σε ποιο δωμάτιο και τι κάνει τη συγκεκριμένη τιμή. Συνεπώ, η ένταση μεταξύ περιβαλλοντική απόδοση και αποτελεσματική προστασία του ιδιωτικού απορρίτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τι δραστηριότητε συντονισμού που επιτρέπουν τη διατήρηση της συνοχής ε, του ρυθμιστικού πακέτου μας. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι πολλά από αυτά που θεωρούμε δεδομένα σε σχέση με το ιδιωτικό απόρριτο και που χαρακτηρίζουν τους κανονισμούς μας έρχονται από εποχές όπου τα πράγματα που κάναμε online ήταν λίγα. Ήταν εύκολα ε, καθοριζόμενα. Είχαμε κανόνες που διέπουν την επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων. Αλλά ας πούμε δεν καλύπτουν την από δημιουργία ε, περιεχομένου στο ίντερνετ από πολλά άτομα όταν εγώ στέλνω ένα μήνυμα σε εσά, ναι, υπάρχει το απόρριτο, αλλά όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών ατόμων και αυτή η αλληλεπίδραση είναι σημαντική, επίσης και οι στάσεις ε, προς, ε, σε σχέση με το απόρριτο έχει αλλάξει επειδή οι πληροφορίε είναι εικονικέ ε, στο διαδίκτυο και μπορώ να αλλάξω διευθύνση email όποτε θέλω, μπορεί να μην με ανησυχούν ιδιαίτερα τα αιτήματα του κράτου να, να με αναζητήσει με τον Google αλλά άλλοι παίρνουν αυτά τα ζητήματα πολύ στα σοβαρά θα πρέπει να το σκεφτούμε όλο αυτό Ίσως χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανονισμούς για ειδικές περιπτώσεις που περιλαμβάνουν παιδιά ή κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο σε άλλες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να μειώσουμε τους κανονισμούς και να αφήσουμε πράγματα που αυτοοργανώνονται από μόνα τους, όπως εμπορεύσουμε δικαιώματα απορρίτου, εφόσον συμμορφώνονται με βασικές αρχές. Και το τελευταίο είναι ότι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που κάναμε τη μελέτη, υποψιάζόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες μορφές πληροφοριών online. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να συμβεί είναι ότι μπορεί σε ένα τομέα διαδικτύου μπορεί να έχουμε βελτιωμένου μηχανισμού επιτήρηση τη συμμόρφωση. Με άλλα λόγια, μπορεί να είναι δυνατόν να ανοιχνεύσουμε, να εχνηλατήσουμε την πρόσβαση σε πληροφορίε. Όταν εσεί μου δίνετε έλεγχο των προσωπικών μου ε, πληροφοριών online, εγώ δεν έχω κανένα, καμία εχνηλάτηση του τι γίνεται με αυτέ τι πληροφορίε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να απαγορεύσω τη διαβίβασή του. Μπορεί να είναι επαρκέ με το, έργο, με το πρόγραμμα Nebula, μια νέα αρχιτεκτονική στι Ηνωμένε το οικιακό κέντρο δεδομένων σας, δεδομένων σας ελέγχει το τι συμβαίνει στα, στα δεδομένα σας. Το τελευταίο σύνολο συστάσεων έχει να κάνει με την αλλαγή που υφίσταται ο κόσμος εδώ. Η διένεξη μεταξύ καινοτομίας και απορρίτου γίνεται σημαντική. Υπήρξε ένα άρθρο για τον Μάρκ Τζούκερμπερ στο γερμανικό τύπο, όπου αναφέρθηκε ότι στη Γερμανία μια μικρή νοσίστατη επιχείρηση που έχει να κάνει με. Ε, δεν θα είχε μπορέσει ποτέ να ξεκινήσει την επιχείρησή του Τζούκερμπερ. Σε ορισμένε περιπτώσει πρέπει πρώτα να περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα πριν να αποφασίσουμε για τη μορφή προστασία που θα επιβάλλουμε. Σε άλλε περιπτώσει θα αναφέρουμε σαφώ του φραγμού, τους κανόνες που δεν θα πρέπει να παραβιάζονται. Ο συνδυασμό ηγεσία και προσαρμοστικότητας είναι πιστεύω η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη. Το απόρριτο είναι ένας τρόπος κλεισίματος των πραγμάτων αλλά μπορεί να βοηθήσει σε έμπιστα περιβάλλοντα όπου έχουμε ιδιωτικό απόρριτα το οποίο μας επιτρέπει να μοιραστούμε ιδέες και όχι να τις κοινοποιήσουμε. Και οι ειδικέ αυτές να είναι δικές μας ιδιοκτησίες. Αυτό είναι αυτά που συμβαίνουν στο διαδικτύο. Θα ήταν δυστυχές αν η ανταπόκριση μα στα σημερινά διαδικτυακά προβλήματα ε, δημιουργούσε πρόβλημα σε ε, χρήστες που χρειάζονται προστασία και τους εμπόδιζε από, το, από πιο ενεργή συνεργασία ή μας εμπόδιζε από το να αναπτύξουμε εναλλακτικέ λύσεις όπως δημόσια κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται για το απόρριτο. Τέλος, ε, θεωρούμε ότι οι σχέσεις ε, που στηρίζουν το ιδιωτικό απόρριτο σε αυτό τον τομέα βρίσκονται σε συνεχείς αλλαγές. Η μεγάλη παροχή υπηρεσιών ίντερνετ Ξέρω ότι έχετε μιλήσει εδώ για το η συνθήκη άκτα, αλλά δεν θα σας μιλήσω εγώ για αυτή. Αλλά τα συμφέροντα του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να εξελίσσονται λόγω της ανάδυσης νέων τεχνολογιών. Ορισμένα πράγματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσω και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα λάβετε αντίγραφα της παρουσίασης και στην τελευταία σελίδα της παρουσίασης θα βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για εμάς και για τους ε, υπευθύνους του Κοινοβουλίου. Ε, ωραία, ακούσαμε τους δύο ε, συντάκτες. Θα ήθελε κάποιος να απευθύνει κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Dostęp do danych osobowych... Και πέστε μα κάτι όσον αφορά την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό συνδέεται με απώλεια του ιδιωτικού απορρίτου. Και συχνά αναδείτε το ερώτημα. Σε ποιο βαθμό η πρόσβαση αυτή είναι επικίνδυνη η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πολύ. Και αυτό ίσως σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε προστασία, να εμποδίζουμε την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Μπορεί και να αποκλέψει τα email κάποιου αλλά επίσης στο ίντερνετ υπάρχουν και προσωπικά οικονομικά δεδομένα, ας πούμε ε, τραπεζικά στοιχεία κάποιου. Μπορούς, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα, αυτές, οικονομικά στοιχεία, τα τραπεζικά, δεν θα διαρρέουν Επομένω, να μην υπάρχει πρόσβαση ούτε στου λογαριασμού μα, ούτε σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ούτε, ούτε και από τραπεζικά ιδρύματα. Για πετε μα, είναι δυνατόν να υπάρχει προστασία αυτών των τραπεζικών δεδομένων. Και να μην μπορεί ο κόσμος να υποκλέψει και χρησιμοποιήσει τα δεδομένα κάποιο άλλο. Να προστατεύεται επομένω και ο λογαριασμό μα και βεβαίω να μην πηγαίνουν τα στοιχεία μα στι διαφημιστικέ εταιρείε. Σε ποιο βαθμό μας μπορούμε να προστατεύσουμε το δυτικό απόρριτο, σε ποιο βαθμό μπορούμε να είναι ασφαλή τα στοιχεία μας. συγκρίνεται τώρα με κάποια άλλα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με, με, με, με κάποιες ε, πολύ ειδικέ περιοχές γνώση, εμπειρογνωμοσύνης όπω α πούμε στατιωτικέ πληροφορίε, πληροφορίε, εξωτερική πολιτική, γιατί και, και πληροφορίε πληροφορίες διακινούνται στο διαδίκτυο. Πολλέ φορέ ε, α πούμε έχουμε και τι ε, κατοικίε. και ε, γίνεται κάποιο συζήτηση με το, το Ιντερνετ, οπότε ε, στέλνονται διευθύνσει παντού. Επομένω, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται αυτά τα δεδομένα. Well, thank you very much for... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, Πρόεδρε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση. Ας ακούσουμε κάποιες τελευταίες σκέψεις από τους ε, συντάξεις. Έχουν ο καθένας 7 λεπτά στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσει. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που πήρα το λόγο μόνο μου. Ε, Αφηρημένο ήμουν. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Προσπαθούμε στην μελέτη να επισημάνουμε το τι συμβαίνει. Προσπαθούμε επίσης όλα αυτά να τα εντάξουμε σε κάποιο πολιτικό πλαίσιο, κοινωνικό πλαίσιο με υπευθυνότητα, γιατί πολλοί τη σήμερα έχουν αυτά τα ερωτήματα και απορίες. Να σας πω επομένως πώς τα βλέπω όσον αφορά την τεχνολογική πλευρά του θέματος σε σχέση με το τι, τι πρακτική ακολουθείται από τις εταιρείε. Ε, ο καθηγητής και θα με συμπληρώσει ε, θα σας πει τα θέματα τα πιο θεσμικά, τα πιο κανονιστικά. Είναι ένα θέμα διαφάνειας. Τι διαφάνεια έχουμε σήμερα. Τι γίνεται με τον έλεγχο, τι γίνεται με τη συνένεση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την νομοθεσία Πρόστασία του ιδιωτικού απορρίτου. Πάντω αυτό το οποίο επισημαίνεται στην μελέτη είναι ότι αν δείτε τι γίνεται σήμερα θα δείτε ότι υπάρχει κάποια βασική ε, δραστηριότητα κορμού α την πούμε που ε, έρχεται σε σύγκρουση κατά κάποιο τρόπο με, την, ε, με τον έλεγχο τα πράγματα γίνονται πιο διάφανα για τις εταιρείε, αλλά ο τρόπος που οι εταιρείε διαχειρίζονται αυτά τα στοιχεία γίνεται όλο ένα και ε, πιο προβληματικό για τα πρόσωπα. Έχουμε επίση τη λεγόμενη διτή ή διπλή διαφάνεια. Ισχύει μόνο και για τις δύο πλευρές. Και υπάρχει έλεγχος και από πλευράς πολιτών οι οποίοι μπορούν να διαπιστώσουν τι απογίνονται τα δεδομένα τους. Διαπιστώνται επίση ότι ε, υπάρχουν θέσει τη αγορά όπου Εκεί δεν μπούμε στις ε, αλλά αν δείτε εκεί τι γίνεται όσον αφορά την ε, αποθήκευση ε, προσωπικών δεδομένων, εκεί υπάρχει μια αρχιτεκτονική σημάδων πληροφορική, όπου κάποιες οργανώσεις ξεβρίσκουν κάποιες λύσεις για το ότι και, και, τελικά αυτές οι λύσεις κατατείνουν στο να υπάρχουν τα δεδομένα και διαθέσιμα για όλους. Άρα, σε μία σειρά χωρών διαπιστώνεται ότι αυτές οι εταιρείε έχουν ε, κάποιο είδους ε, επαγγελματική ηθική, επαγγελματική πρακτική που είναι εναλλακτική σε σχέση με την παραδοσιακή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από τη δική μου χώρα, την Ολλανδία. Ε, όμως αυτές είναι συγκεκριμένοι παίκτε στην αγορά, συγκεκριμένες θέσει στην αγορά και τώρα από πλευρά πολιτική, το πώ μπορεί κανεί ε, να, να δει τι γίνεται στην ε, κυρίως αγορά. Είναι πολιτικό πολύ το θέμα. Πια θα σας τα πει ο συνάδελφος, αλλά ε, είναι θέμα καρότου και ραβδιού. Πώς είναι το καρότο και πώς είναι το ραβδί. Να υπάρχουν τέτοιου είδους ε, υποδομές, τόσο ώστε να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα. Να έρχεται κανείς σε επαφή σε αυτούς που πάνε να, να αυτά τα στοιχεία. Οπότε ε, αυτό που έχει σημασία είναι να έχουν όλες τις πληροφορίες και οπότε πια τα πράγματα δυσκολεύουν και θα πρέπει πια κανείς να είναι βέβαιος ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πάρει το δεδομένο. Η ιδέα κυβερνική πρακτική Ε, μπορεί να γίνει πρωτοπόρα και να εξασφαλίσει ότι αυτές οι πρακτικές είναι ανοιχτέ και αποτελούν ευκαιρία για μια νέα κουλτούρα. Πολλές φορές επομένως κάποιοι υπάρχουν υπηρεσίες, δεν είναι αυτές οι υπηρεσίες στο επίπεδο που θα προσδοκούσε κανείς. Επίσης, πάρα πολλά συμβάντα, γεγονότα, περιστατικά δείχνουν ότι το επίπεδο της προστασίας αφήνει περιθώρια να κάνει κανείς μέσα από ένα σύστημα κάποιες ε, κινήσεις που δεν θέλει να κάνει το κάθε φυσικό πρόσωπο το ίδιο. Αυτό γίνεται με προγραμματισμό. Είναι αυτό δυνατό χωρίς να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας οδηγεί σε κάποιο είδους υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά και με περιθώριο του να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας. Υπάρχει μια συνάδελφο που θέλει να κάνει μια ερώτηση, οπότε θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα της επιτρέψουμε να την κάνει τώρα, ώστε να μπορέσει να απαντήσει ο καθηγητής. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση. Αναρωτιόμουν η υπεύθυνη της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της ε, βρήκατε κάποια συγκεκριμένα μοτίβα καινοτομίας το καινοτόμα ε, στην Ευρώπη σε σχέση με τις αμερικανικές επιχειρήσεις δεδομένων των διαφορετικών νομοθεσιών απορρίτου που έχουμε στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ποιες διαφορές είναι αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Υπήρχαν κάποιες διαφορές Ορισμένες από τις διαφορές αφορούν το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ίντερνετ Πρέπει να πούμε ότι ο τομέας του διαδικτύου βλέπει την Ευρώπη να έχει μείνει πίσω σε θέματα καινοτομία, όχι μόνο όσον αφορά το απόρριτο, για διάφορους λόγους που είμαι βέβαιος ότι όλοι κατανοούμε και διαρκώ ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Επίσης, ωστόσο, αληθεύει ότι η υποκείμενη δομή εμπιστοσύνης, οι νομικές απαιτήσεις ε, οδηγούν αυτή τη διαφορά ως εξής. Ο βαθμός στον οποίο οι δημόσιες αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο εμπιστοσύνη ε, και συνεπώς ε, μπορούν να παραβιάσουν το απόρριτο είναι πολύ διαφορετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό οι άνθρωποι να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα και την αντιστήξη δεδομένων, συνδυασμό διαφέρων ε, δεδομένων μεταξύ ατόμων. Αυτό είναι κάτι νόμιμο. Μπορεί να το κάνει νόμιμα ο δημόσιος τομέας. Ταυτόχρονα, μία από τι καινοτομίε είναι ότι δίνουν οι κυβερνήσει πολλέ από τι δραστηριότητέ του σε ε, εταιρείε του ιδιωτικού τομέα. Εδώ λοιπόν να μιλάμε για μια καινοτομία που μπορεί να πλήξει το ιδιωτικό απόρριτο. Όταν ιδιωτικοποιούμε πράγματα τα οποία βρίσκονται στη σφαίρα της δημόσιας εμπιστοσύνης από την άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου υπάρχει μικρότερη εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και μεγαλύτερη προς τις επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επειδή διάφορα περιστατικά έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε σχέση με το απόρριτο, παρατηρήθηκαν πολλές πρωτοβουλίες βελτίωσης της ευθύνης όσον αφορά το απόρριτο για διάφορες εταιρείε παροχής ίντερνετ που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και ισχυρές πολιτικές και ιδιωτικού τομεί όπως τη World Gardens όπου το ιδιωτικό απόρριτο ενό ατόμου διασφαλίζεται χάρη στον περιορισμό των ανθρώπων που μπορούν να έχουν προσβάσει τα δεδομένα σα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτε έχουν δείξει ότι η προστασία που παρέχουν αυτές οι πολιτικές είναι αντιστρόφως ανάλογη με το να αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Πολύ προφανείς λοιπόν επιλογές απορρίτου με πολύ μικρή προσπάθεια εφαρμογής αυτών των επιλογών. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε λειτουργική επιχειρησιακή καινοτομία στην Ευρώπη και εδώ μιλάμε όχι μόνο για τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και οι μηχανισμοί αναζήτησης ε, που σέβονται τα... το ιδιωτικό απόρριτο είναι ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο δεν αφορά συγκεκριμένα τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά αποτυπώνει έναν τομέα όπου η καινοτομία είναι αρκετά έντονη και βασίζεται στην προηγούμενη ερώτηση. Ένας τομέας ε, ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδομένων και όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι τα ηλεκτρονικά αρχεία, ιατρικά αρχεία ασθενών. Είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς ε, συνένεση, ειδικότερα εάν είναι ε, ισχυρά ασθενή στι Ηνωμένε υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που ελέγχει τη συλλογή δεδομένων, ηλεκτρονικών δεδομένων και ιατρικών αρχείων ασθενών. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Διένεξη συμφερόντων θα έλεγα. Όταν έχουμε ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών που δεν μπορούν να τα δουν άλλοι γιατροί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραπέμψουμε τους ασθενείς στη σωστή φροντίδα στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου οι ασφαλιστικές τελείες παίζουν τεράστιο ρόλο, η πρόσβαση στις, ε, ε, στα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία αυτών των συστημάτων προστασίας του ιδιωτικού απορρίτου. Εάν εγώ ως γιατρός γράψω τα πάντα ως, για εσάς ως ε, ασθενή, υπάρχει κίνδυνος να σας χάσω προς όφελος ενός άλλου. εάν δεν τα γράψω όλα, τότε δεν έχω αναλάβει τις ευθύνες μου ως γιατρός. Ε, αν γράψω ακριβώς αυτές τις πληροφορίες που μπορεί κάποιος άλλος γιατρός να χρειαστεί για να σας θεραπεύσει, εδώ έχουμε έναν τομέα όπου η προστασία του ιδιωτικού απορρίτου ε, ε λειτουργεί ως μπούμεραγκ με τους κανόνες του ανταγωνισμού. όταν ε, οδηγούμε τους ανθρώπους για ατομική προστασία τους ε, έχουμε ας πούμε το παράδειγμα του phishing σας δίνουν έλεγχο των δεδομένων σας αλλά ποιος σας προστατεύει από αυτούς που προσπαθούν να ελέγξουν εσάς ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ευρώπη έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτόν τον τομέα παραμένουμε άνθρωποι Ωραία, ευχαριστούμε τον καθηγητή Κέιβ και τον κύριο Λίσχαουτ για την παρουσίασή τους, αυτής της μελέτης τους, ενημερωτικά για τις ε, πληροφορίες και τις γνώσεις που μας διέθεσαν. Τους ευχαριστούμε και έτσι ολοκληρώνεται η παρουσίαση του, ε, της εργασίας σας για την Ήτρα. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, Σύγκρινε τώρα τις εργασίες μας και έχουμε τώρα ε, μια εισήγηση. Παρακαλώ να βγει όποιος δεν ενδιαφέρεται για το, τις υπόλοιπες ε, συζητήσεις που θα κάνουμε. Είναι μαζί μας λοιπόν, ο πρόεδρος, ο καθηγητής Ποτόσνικ. Ο καθηγητής Ποτόσνικ, ο οποίος είναι διευθυντής του ACER στα αγγλικά, Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αργών Ενεργείας. θα κάνει μια σύγχυση 20 λεπτών. Και ε, τον ε, Ιούλιο, πέρσι τα είχαμε ξαναπεί στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει στα Ιταλικά ο κ. γιατί μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να σας παρουσιάσω τις ε, δραστηριότητες του οργανισμού μας και με την αδειά σας θα συνεχίσω την εισήγησή μου ή στα αγγλικά. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ τις δραστηριότητες του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας. Την τελευταία φορά που τα έχαμε ξαναπεί ε, ήταν τον ε, Ιούλιο του 2011 σε μια παρόμοια ε, ευκαιρία. Τώρα θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη για τον συνάδελφο τον κύριο Μπόλτς ο οποίος είχε προσκληθεί αλλά τελικά είχε κάποιο πρόβλημα και δεν μπόρεσε να παραστεί. Πέρσι όταν ήμουν εδώ, σας είχα πει ότι προσλαμβάνουμε προσωπικό για τον οργανισμό μας. Και είχαμε πει ότι η διαδικασία προσλήψεων πρόκειται να τελειώσει πέρα του έτους. Ε, προσλαμβάνουμε αυτούς που προβλέπουν στο καταστατικό μας. Επίσης, ολοκληρώσαμε τους διορισμούς. Ε, έχουμε επίσης και κάποιο ε, όργανο προσφυγών ε, αυτό ε, τον Δεκέμβριο ε, κατά την πρώτη συνεδρία. Σε πάση τώρα είμαστε πλήρως λειτουργικοί από πάσα άποψη. Όμως, ακόμα, ακόμα δεν λειτουργούμε με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, διότι από τότε που ξεκίνησε η υπηρεσία μας έχουμε επιπλέον αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν σε σχέση με την αγορά, σε σχέση με τη διαφάνεια. 28-12 ε, τέλο πάντων θεσμικά μας ανατέθηκαν αυτά τα νέα καθήκοντα. Επίσης μας έδωσαν επιπλέον ε, αρμοδιότητες δυνάμει του κανονισμού που αφορά τις κατευθυντήριες για τα διευρωπαϊκά ευρωπαϊκά, με τα διευρωπαϊκά συγγνώμη, ενεργειακά δίκτυα και τη σχετική υποδομή. Αυτά και οπότε έτσι ε, θα σας πω για το τι γίνεται, ε, τι ισχύει ε, σήμερα κατόπιν αυτών των αλλαγών. Πάντως με την ευκαιρία να ε, ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, διότι χωρίς διακοπή μας στηρίζει ε, κατά όλη μας την πορεία και όσον αφορά τη διαδικασία θέσπισης αυτού του τελευταίου νομοθετήματος για τις ομοριτές μας. Η αρχική μας εντολή καταρχήν αφορούσε την ε, ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς ή αγορών και άρα οι βασικές μας δραστηριότητε, σύμφωνα με το καταστατικό αφορούν ε, το πρόγραμμα το 10 για τα δίκτυα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό ε, στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτών των δικτύων Οπότε έτσι θα βρούμε και την ε, ε, αφετηρία για κάποια προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος από ό,τι φαίνεται αυτή την ε, διάσταση τα πράγματα, κατά τη γνώμη μας, οπότε και γι' αυτό θεωρούμε ότι στο όλο παζλ αυτό θα είναι σημαντικό. Επίσης έχουμε αυτούς τους πρώτους 15 μήνες θα έχουμε το τρίτο πακέτο και κάποιους κώδικες που προβλέπει κοινού κανόνες που πρόκειται να θεσπιστούν για τις ευρωπαϊκές ε, ενεργικές αγορές. Επομένω, θα έχουμε κοινού τέτοιου κανόνες και όχι απλή εναρμόνιση. Θα σας πω περισσότερες ε, λεπτομέρειες σε λίγο. Πάντως, αυτό το οποίο προωθούμε είναι τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας γιατί βεβαίω ε, χρειάζεται να υπάρχει υποπτία και έλεγχος κάτι το οποίο η εντολή μας το αναβάθμισε. Με δύο λόγια τώρα. Τι έγινε τους τελευταίους 15 ε, με 18 μήνες. Είχαμε αυτά τα προγράμματα, τα τρία και το τέταρτο τώρα που προβλέπεται για αυτό το καλοκαίρι, ε, τα οποία ε, τα προχωρούμε και ολοκληρώνουμε τώρα για αυτό το πρόγραμμα του Θέρους το, τη διαδικασία της ε, διαβούλευσης και αυτά θα είναι, αυτοί θα είναι οι, οι κώδικες δικτύων για την αγορά ε, των ε, ε του, του ηλεκτρισμού και θα τα πούμε ε, το τι έγινε όταν ξαναρθούμε του χρόνου. Έχουμε δύο κατευθυντήριες όσον αφορά το φυσικό αέριο και τώρα ολοκληρώνουμε μια τρίτη κατευθυντήρια για την ανταλλαγή των δεδομένων και ήδη έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε και ένα τέταρτο. Οπότε συνολικά ε, περί τα τέλη του έτους ε, θα έχουμε προγραμματίσει να έχουμε 8 και 4 κατευθυντήριες πλαίσια που θεωρούμε ότι θα είναι η σπονδυλική στήλη ε, για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης, ε, δεν θέλω να επιστρέψω στις λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να σας να σταθώ και σε άλλα δύο θέματα πρώτα-πρώτα. Η γνωμοδότηση όσον αφορά αυτό το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου, τα είπαμε πέρσι και τονίσαμε τι γίνεται και θα υπάρξει επίσης μια γνωμοδότηση που θα αφορά το, την αγορά του ηλεκτρισμού γιατί βεβαίως ε, ε, αποφασίστηκε κάποια τέτοια παράλληλη πορεία. Για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο δεκαετές πρόγραμμα. Πρόκειται για κάτι το νέο και για πρώτη φορά επομένω έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή ε, σημαντική ε, διάσταση σε, αυτή, σε αυτόν τον δεκαετή προγραμματισμό και εμεί ε, θέλουμε ακριβώ αυτές τις ε, διαδικασίες να τις προσέξουμε. Τώρα να σας τονίσω κάτι άλλο τελευταίο αφορά κάποια σύσταση πρώτη η οποία εξεδόθηκε με δική μας ε, πρωτοβουλία όσον αφορά αυτά τα οικονομικά δικαιώματα διάδοσης, μετάδοσης ε, πρόκειται για ε, κάποια, κάποιες διατάξεις που δεν, δεν υπάγονται στον ε, δημοσιονομικό γενικό κανονισμό είναι ειδικέ ρυθμίσεις για τον ενεργειακό τομέα. Τώρα πάμε στο θέμα της εντολής μας για το οποίο θέμα ξέρετε εσείς περισσότερα από ό,τι εγώ, μια που τώρα πρόσφατα ασχοληθήκατε. Άρχισε η εντολή μας επομένω τον Δεκέμβριο πέρσι. Κάποιες από τις σχετικές διατάξεις ευθύς αμέσως ήταν εφαρμοστέας, ε, υπήρχαν όμως ε, είχαμε κάποιες διατάξεις για παραβίαση του καθήκοντος εμπιστοσύνη, insider trading και επίσης ε, και επίσης και για παραβίαση των ε, κανόνων ανταγωνισμού και κατάξει δεσποζούσης θέσεως και επίσης είπαμε ότι έχουμε κάποια άλλα θέματα κατάρτισης και κάποιες ε, άλλες ρυθμίσεις που θα αφορούσαν καταγγελία σε περίπτωση παραβάσεων. Και όλα αυτά σας τα τονίζω διότι για αυτά τα δύο θέματα, για αυτά τα θέματα έπρεπε να έχουμε κάποιο είδους υποστήριξη κάποιο είδου ε, κατάρτιση να υπάρξει ευθύ εξ αρχή. Και έχουμε ε, και κάποια προθεσμία, η οποία θα εκπνεύσει κατά τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει ο οργανισμό μα να δημοσιεύσει το σχήμα ε, μεταφοράς δεδομένων από τα εθνικά προς το ευρωπαϊκό μητρό, το οποίο είναι κάτι το νέο, το οποίο προσετέθη εκ των υστέρων κατά τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Οπότε και ασχολούμαστε τώρα με αυτό αργότερα. Ανάλογα με, την, με το timing της εφαρμογής ξεκινήσαμε με καταγραφή των όσων συμμετέχουν στην αγορά και στη συνέχεια είπαμε θα έχουμε και ένα σύστημα εποπτείας ελέγχου για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε. Να, σα δείχνω τώρα τι έχουμε κάνει, δεν μπορώ να μπω τώρα στι λεπτομέρειε. Έχετε πάρει τα σχετικά έγγραφα. Είναι μια απλή απαρίθμηση περιστατικών. 29 Ιουνίου η τελευταία ημερομηνία, όχι 28 Δεκεμβρίου. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε αυτού του είδους το σχήμα δεδομένων για τους συμμετέχοντες στην αγορά. εμπειρίες επομένως ε, δημοσιεύτηκαν κατά τα τέλη του προηγουμένου έτους ε, κατόπιν ε, το που προβλέπει η εντολή μας. Δεν μπορούμε να είμαστε δεσμευτικοί σε αυτές μας κατευθυντήριες, απλώς απευθυνόμεθα προς τις ρυθμιστικές εθνικές αρχές, αλλά πάντως ο κλάδος θεωρεί ότι αυτά που λέμε αποτελούν σημείο αναφοράς. Για κοιτάξτε τώρα τι λέει παρακάτω όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα κάνουμε το επόμενο 1,5 χρόνο. Ε, this work will be completed. Και μπορείτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους. Και ε, θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με, του, με αυτούς που διαχειριζόνται κάποια συστήματα, τους σύστημα περίπτωσης και σχεδόν για τους κώδικες ε, ή κωδικούς δικτύων έχουμε ολοκληρώσει. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό για να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014 η αγορά ενέργειας. Σήμερα επεξεργαζόμαστε αυτούς τους κωδικούς για το φυσικό έργο. Και έχουμε άλλους 12 να επεξεργαστούμε. Αυτό θα είναι το κύριο έργο μας για τον επόμενο 1,5 χρόνο. Να έχουμε επίση και μια αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Και να δούμε μέσω της επιτροπολογίας πώς θα τα κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτικούς νομικά κανόνες για την αγορά ενέργειας. Ήδη στόχοι των αγορά φυσικού αερίου έχουν μπει στο πρόγραμμά μας και σιγά σιγά προχωρούμε και για τον ηλεκτρισμό και εκεί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα ζητήματα. Άλλωστε, προσπαθούμε να σταθμίσουμε, τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γνωμοδοτήσει επίση όσον αφορά αυτό το δεκαετέ πλαίσιο, πρώτα πρώτα για τον πληθυσμό και του χρόνου για το φυσικό αέριο. Όχι όπω προανέφερα, ταυτόχρονα η διαδικασία οι διαδικασίες πρόκειται να ενοποιηθούν, πρόκειται να, να συγκλίνουν και για τις δύο αγορές αερίου και ηλεκτρισμού. Τώρα, έχουμε κάποιε αρμοδιότητε ελεγκτικέ. Αυτό το προβλεπόταν από το ιδρυτικό καταστατικό και τον σχετικό κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά, για, για την τιμολογιακή πολιτική και για την τήρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Όπως προανέφερα, ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση της εντολής ε, και ουσιαστικά πολύ πριν αρχίσει να ισχύει το σχετικό νομοθέτημα. Και πέραν τώρα αυτού του σχήματος καταγραφής το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τώρα και μέχρι την επόμενη χρονιά θα φροντίσουμε για την εκτέλεση της εντολής επομένως άμεσα αυτό θα μας απασχολήσει θα είναι το πώς θα προτείνουμε κάποιες συστάσεις για τις, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την ρύθμιση των συναλλαγών όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, εκείνα τα οποία υπόκεινται σε εμπορία στην Ευρώπη. Επίσης θα αναπτύξουμε κάποια μεθοδολογία ελέγχου. Στη δε συνέχεια θα ξεκινήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Μητρό και κάποιες μεθοδολογίες ελέγχου. Και να, με τι προσέγγιση θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο, συλλογή δεδομένων, ε, ανάλυση αυτών. Βλέπετε εδώ αυτά τα κυτρινοπά κουτάκια, τα τρία που είναι στη σειρά διαγώνια. 500.000 τέτοιες συναλλαγές ή δεδομένα θα έχουμε την ημέρα αυτοματοποιημένος έλεγχος θα γίνεται και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε πού έχουμε περιστατικά ή δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν κάποια αντικανονικότητα αν αφορούν πρόσωπα θα αναφερθούμε σε αυτά ιδάλλως θα απευθυνθούμε στις εθνικές ελληνικές αρχές και τώρα Για να δούμε τώρα τι θα γίνει όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τα έργα υποδομή με αυτόν τον κανονισμό ο οποίος αναμένεται να αρχίσει να ισχύει αρχάς επομένου έτους εκεί θέλουμε να γίνει κάποια επισήμανση των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ανάλυση κόστους-οφέλους ε, σε και σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό σε δεύτερη φάση επίπεδο, κάτι το οποίο θα γίνει μεταξύ τέλους του ενωστότους και, μετα, και μέχρι τον Ιανουάριο του επομένου. Επίσης θα μας δηθεί και γνωμοδότηση όσον αφορά τη μεθοδολογία κόστους ε, ωφέλους για, του, για, operators των συστημάτων μετάδοσης, ε, κίνητρα, πώ οι επιπλέον κίνδυνοι θα σταθμίζονται. Να, επομένω, τι περιμένουμε να γίνει τον επόμενο 1,5 χρόνο. Το δε πρόγραμμα εργασία για του χρόνου θα αρχίσει πάρα πολύ σύντομα. Θα το προσφέρω στο Συμβούλιο μα αλλά και στο Κοινοβούλιο του χρόνου. Και έλεγα τώρα στην Πρόεδρο πώς μπορούμε να κάνουμε τον Ιούλιο μία συνάντηση για την να γίνει σχετική παρουσίαση στις Βρυξέλλες. Για να θίξουμε τώρα τα θέματα τα δημοσιονομικά. Έτσι θα ανταποκριθούμε στις σημαντικές προκλήσεις που έχουμε. Διότι βλέπετε ότι αυτός είναι ο προπολογισμό μας τον οποίο έκρινε το Διευθυντικό Συμβούλιο για το χρόνο. Σημαντική αύξηση έχουμε σε δύο βασικά, βασικές κατηγορίες εγκαταστάσεις χρόνο θα πρέπει να πληρώσουμε στη Λιουμπλιά, στη Λιουμπλιάνα τις εγκαταστάσεις μας γιατί μέχρι φέτος οι Σλοβαίνοι ε, βάσει συμφωνία που γίνει μας φιλοξενούν δωρεάν. Επίση έχουμε και το θέμα τη εξεργασίας των δεδομένων που αφορά την υλοποίηση τη εντολή μα. Οπότε ε, θα δείτε τι γίνεται τώρα με αυτέ τι δαπάνε Φτάνουμε τα 12 εκατομμύρια για το χρόνο όσον αφορά την, την, την, την, τις προβλέψεις, αλλά σύμφωνα με το σχέδιο προπολισμού που έκανε η Κομισιόν τον Απρίλιο, η υπηρεσία μας θα έχει διαθέσιμα μόνο 9 εκατομμύρια του χρόνου. There are also challenges um, in the approaches and there are challenges. Και επίσης έχουμε εμ, συγκεκριμένο, συγκεκριμένη πρόβλεψη για το REMIT, το REMIT τέλο πάντων που αφορά το προσωπικό. Αυτό που κάνουμε δεν γίνει πουθενά στον κόσμο. Γιατί υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολύ λίγε προηγούμενε εμπειρίε σε εθνικό επίπεδο, αλλά διεθνώ πάρα πολύ λίγα πράγματα ακόμα και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σιγά σιγά μόλις τώρα κάνουν αυτό το οποίο εμείς ε, προβλέπουμε και υλοποιούμε. Βλέπετε πόσο περίπου τα πράγματα και για κοιτάξτε τι γίνεται με τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εδώ θα πρέπει η υλοποίηση να γίνει πριν αποφασίσουμε για τη μεθοδολογία αξιολόγηση. Τώρα για την επάνδρωση του προσωπικού ο προβλημός προϋπολογισμός βλέπετε τι προβλέπει και έχουμε επίσης και σε σχέση με, το, με τη δέσμη μέτρων για, το, για, τα, για τις υποδομές προβλέπονται επίσης προϋποδότηση και το σχέδιο προς του 2013 δεν καλύπτει όλες τις δαπάνες. Τέλος. Τα τρία εκατομμύρια τα οποία μας λείπουν προσεγγίζουν πάρα πολύ τις επενδύσεις που είπαμε ότι θα μας χρειάζονται για του χρόνου. Επομένως, διακυβεύεται πάρα πολύ η δουλειά μας το 2014. Άρα, αν πάμε λίγο προς τα πίσω, θα δούμε ότι τα περισσότερα θέματα στον προπολογισμό μας δεν διακρίνονται από καμία ελαστικότητα. Δηλαδή το, το, το, το προσωπικό πρέπει, το προσωπικό να πληρώνεται. Τα κτίρια επίση. Και έχουμε 3,4 εκατομμύρια τα οποία σκοπεύουμε να επενδύσουμε του χρόνου. Αλλά τελικά θα έχουμε λιγότερο μισό εκατομμύριο και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο που θα κάναμε ε, με τα 3,5. Οι εθνικές αρχές έχουν βοηθήσει, ναι για να εφαρμόσουμε το REMIT και επίσης ε, τώρα έχουμε ακόμα περισσότερη δημοσιονομική πίεση γιατί έχουμε νέες αρμοδιότητες αλλά και εδώ δυσκολεύονται οι εθνικέ να βοηθήσουν, γιατί όπω ξέρετε υπάρχουν περικοπέ και στου εθνικού προπολογισμού. Τέλο πάντων, πάντοτε υπάρχει φω στην αρχή του τουνέλ. Οι δε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν τώρα ότι θα πρέπει να μα δώσουν περισσότερα χρήματα για το 2013. Ακόμα πρέπει να συνοηθούμε για το πώ θα υλοποιηθεί αυτό. Από ό,τι μου είπαν, μπορεί να γίνει αυτό με εσωτερική μεταφορά πόρων ή με επιπλέον αίτημα προ τι δημοσιονομικέ αρχέ. Τέλο πάντων, ό,τι για να κάνουμε θα πρέπει να γίνει αμελητή. Σα διαβιώνω πάντω ότι ό,τι και να γίνει ο οργανισμός μας, το Acer, θα, κάνει, θα αξιοποιεί όσο μπορεί περισσότερο και καλύτερα τους πόρους που του και σας ευχαριστώ και συγγνώμη που με Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο ε, Ποτροσκή. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τον συνεπαρακαλώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Δ. Αποτόσνικ, για την παρουσίασή σας. Δυστυχώς τα αντίτυπα των διαφανειών εγώ έλαβα μόνο μερικά από τα αντίτυπα. Κατά κάποιο τρόπο θα ήθελα να έχω και τα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι μιλάμε εδώ για ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δομή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε αυτούς τους οργανισμούς ώστε πραγματικά να είναι ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκοί. Αναφέρομαι στο ηλεκτρικά δίκτυα, αλλά όχι μόνο. Κατά μέρα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό, διότι ειδικότερα αυτό το επίπεδο, ειδικότερα με την ε, δημιουργία μιας βάσης υψηλής ε, απόδοσης για τις μεταφορές ε, με διαρκή επιτήρηση υψηλού επίπεδου θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ηλεκτρισμού ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας γενικότερα. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα, ωστόσο πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή η προσέγγιση με αυτόν τον οργανισμό που συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές μπορεί να παρέχει αυτές τις εγγυήσει ευρωπαϊκής λειτουργίας πραγματικά αποτελεσματικής και για το δίκτυο φυσικού αορίου υπάρχουν ανάλογα προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές αποθήκευσης. Και εδώ είμαστε εμείς ή όχι, διότι αυτό αφορά την γενικότερη απόδοση. Αναφέρομαι δηλαδή ειδικότερα στην αιωλική ενέργεια που πάντοτε θεωρείται υπερβολικά πολυπίκυλη. Αλλά αν έχουμε αυτή τη βάση που αφορά ολόκληρες τις πηγές αιωλικής ενέργειας και υπάρχει μια καταγραφή των ε, χώρων όπου δραστηριοποιούνται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά την υδροελεκτρική ενέργεια και να συμπληρώσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά την ε, ηλεκτρική ενέργεια για την υποστήριξη της αιωλικής και να πράξουμε γενικότερα όλα αυτά βάσει αυτής της οπτικής. Με αυτή μια τέτοια προσέγγιση ε, την έχουμε ή πρέπει να αναμένουμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε τον συναδέλφο κύριο Πρόντι, το λόγο έχει η κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε κυριε ποτορσνικ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας που μας δείχνει πόση δουλειά απαιτείται για τα σχετικά σύντομα πολιτικά έγγραφά μας. Σε συγχαρητήρια λοιπόν για τη δουλειά που έχετε κάνει. Χαίρομαι πολύ που ακούω ότι δημιουργήθηκε επιτυχώς ο οργανισμός ε, χωρίς ε, προβλήματα όσον αφορά το προσωπικό. Με, ένα, σημαντικό πρόβλημα όμως ε, τον προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πάντα ήταν ε, υπέρ της ε, αγοράς ενέργειας και πιστεύω ότι είναι ευθύνη μας ε, να ενδυναμώσουμε όλους τους οργανισμούς ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους σύμφωνα με την νομοθεσία μας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εφαρμοστεί το REMIT σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που μας υποδείξατε τρόπους να λύσουμε το θέμα αυτό. Μήπως ε, μπορείτε να σχολιάσετε περαιτέρω το θέμα αυτό. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή βρίσκονται όλα πια στα χέρια τα δικά σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να κλείσει επιτυχώς το θέμα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν δεν βρούμε λύση, ποιος είναι ο κίνδυνος. Διότι η διαφορά στο προϋπολογισμό είναι αρκετά σημαντική. Θα ήθελα επίσης ε, να σας θέσω άλλη μια ερώτηση σχετικά με την απελευθέρωση της ε, αγοράς ενέργειας. Υπάρχει απόφαση ότι θα πρέπει να ε, πραγματοποιηθεί ε, αυτό το 2014, αλλά ήθελα να ρωτήσω, τι, θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας, πώς προχωράνε τα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. <laughs> Euh, Δίνω το λόγο, το λόγο στον συνάδελφο Βαλσίτης και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ρόδε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. αναφέρατε μια σειρά προβλημάτων, κύριε Διευθύντα, που αντιμετωπίζετε σήμερα. Καταλαβαίνω την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε. Αναφέρατε επίσης ε, ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό ε, ε, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι Βεβαίως ότι κάποιοι ειδικά από την ε, Ανατολή θα πλήρωναν ακόμα περισσότερα για να, για να μην κάνετε τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να πιέσουμε την Επιτροπή ώστε να δεσμευτεί και να μπορείτε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Εάν ε, δεν έχετε το απαραίτητο λογισμικό και τον ε, απαραίτητο εξοπλισμό, η δουλειά σας θα είναι μάταιη. Στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει, συζητάμε ίσως εδώ και τρία χρόνια την ανάγκη δημιουργίας ε, της ενιαίας αγοράς, αλλά όσον αφορά πρακτικά θέματα, όπως είναι η, ε, διαβίβαση, η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στους τομείς του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου, φαίνεται ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, τα οποία δεν θέλουν να ανταλλάξουν δεδομένα και θέλουν η υποχρεωτική ρήτρα να γίνει προαιρετική. Ε, να έχουμε δηλαδή may αντί για shall στην σχετική διάταξη. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι πολιτικό. Πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν να χάσουν το μονοπόλιο τους, διότι έχουν κάποιες συμφωνίες ε, και συμβάσεις που τους επιτρέπουν να ε, έχουν ρεύμα σε φτηνότερη τιμή. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω απόλυτα τις εργασίες ε, του οργανισμού σας και να σας ενθαρρύνω να δημιουργήσετε κοινούς κανόνες για μια κοινή αγορά ενέργειας. Ε, δεν θα επαναλάβω ε, όλα όσα είπατε τώρα, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στην συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας στα κράτη-μέλη που αναφέρατε εσείς. αναφέρατε ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Πώς μπορεί να λυθεί στο μέλλον ενδεχομένως με κοινέ προσπάθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στο κατάλογο. Σας δίνω λοιπόν, κύριε Ποτόσνικ, απευθείας τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, εξωτήμα μέλη, για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και την ενθάρρυνση και τη στήριξή σας. Όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν είναι πολύ σημαντικά και θα χρειαζόμασταν πολύ χρόνο για να τα συζητήσουμε ικανοποιητικά. Αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια ε, πρώτη σύντομη εικόνα, κατά την απόψή μου φυσικά, προς τον κύριο Πρόντι. Πράγματι, αποτελεί έναν από τους στόχους της ενιαίας αγοράς, της εσωτερικής αγοράς, να ενοποιήσει τις εθνικές αρχές ε, όχι μόνο απόψη κανόνων αλλά και απόψη υποδομών. Σήμερα έχουμε δύο στόχους μπροστά μας το 2014 για την ενοποίηση των αγορών συγγνώμη για την ενοποίηση των κανόνων για τις αγορές και το 2015 για την κατάργηση των ε, νησίδων ενέργειας Ανέφερα ήδη στην παρουσίασή μου ότι ένα από τα κύρια καθήκοντα του οργανισμού είναι να παρέχει γνωμοδότηση για το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα νέο μέσο και όπως ήδη ανέφερα για πρώτη φορά το πρόγραμμα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα δικτύων με ισχυρή εθνική, ευρωπαϊκή διάσταση προγραμματιζόταν μέχρι τώρα σε διμερές επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο σε διμερές το πολύ. Τώρα δίνεται έμφαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι γι' αυτό. Αναφέρατε τουλάχιστον δύο από αυτούς. Η διείσδυση νέων τεχνολογιών σημαίνει ότι θα χρειαστούμε πιο ισχυρά και πιο έξυπνα δικτύα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ήδη σήμερα παρατηρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα χειρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και η κατάσταση θα επιδεινωθεί εκτός εάν υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τους ε, ένσω, συνεργαζόμαστε στενά και επίσης ε, συνεργαζόμαστε στις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και για το νέο πακέτο για τις υποδομές, διότι η ευθυγράμμιση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι υποδομές θα οικοδομηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι ουσιαστική. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα μέχρι σήμερα. Σήμερα έχουμε λοιπόν τα μέσα ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα απομακρυνθούν οι φραγμοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εμείς ε, οι φορείς ε, μετάδοσης, συστημάτων μετάδοσης, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργήσουν όλα αυτά σωστά. Στην κυρία Τζόρνταν, ε, σας ευχαριστώ για την ενθαρρύνσή σας. Ναι, όντως ε, αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση. Όταν συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, ε, το αναγνώρισαν ότι ίσως χρειαστούμε περισσότερους πόρους. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό ε, σε διοικητικές διαδικασίες της Κομισιόν, ειδικότερα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά μου είπαν ότι ένα από τα δύο πιθανώς θα λειτουργήσει. Ε, αν φυσικά θελήσουμε να κάνουμε και άλλη απέτηση από τις αρχές προεπλογισμού θα ήθελα την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής ειδικότερα για το θέμα. Αυτό που διακυβεύεται το REMIT ε, μπορεί ήδη να εφαρμοστεί. Ήδη η απαγόρευση ε, για την εμπορία και την κατάχρηση της αγοράς υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα μέσα για να το πράξουμε. Όταν θα έχουμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να συλλέγουμε, να παρακολουθούμε δεδομένα και να παρακολουθούμε τις αγορές, τότε θα γνωρίζουμε κατά πόσο οι αγορές λειτουργούν τόσο καλά όσο ελπίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το REMIT δεν αποτελεί πρόσθετο κομμάτι, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ενοποίησης. Σε μια ενοποιημένη αγορά η εμπορία θα είναι πιο περιπλοκή και ουσιαστικά αυτό θέλουμε. Θέλουμε περισσότερο διασυνοριακό εμπόριο όταν αυτό είναι αποτελεσματικό. Επιστεύω ότι οι καταναλωτές μας στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν να γνωρίζουν, αξίζει να γνωρίζουν ότι λειτουργεί σωστά και ότι υπάρχει επαρκή ακαιρεότητα και ε, διαφάνεια. Αυτό λοιπόν διακυβεύεται. Το να διασφαλίσουμε ότι η σωστή λειτουργία των αγορών. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όντω η αγορά λειτουργεί σωστά, αλλά δεν μπορώ να σα το εγγυηθώ και αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σα το επικυρώσω. Όσον αφορά την ε, απελευθέρωση για το 2014. στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κλείσουμε και να πάμε διακοπές. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και ορισμένες από τις προκλήσεις που ήδη αναφέρατε θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά το 2014. Οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, το ζήτημα της αηφορία, η πρόκληση της αηφορίας και τη βιωσιμότητα θα υπάρχουν ακόμη για πολλά χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι στόχο για το 2014, τουλάχιστον όπω το έχω καταλάβει εγώ, όπω το έχω ερμηνεύσει εγώ, θα είναι να φροντίσουμε μέχρι τότε η αγορά να λειτουργεί αρκετά καλά. Θα το καταφέρουμε, έτσι πιστεύω. Στον ηλεκτρισμό παρατηρούμε, διαπιστώνουμε μάλλον ότι η παράλληλη υλοποίηση, καθώς αποφασίζονται οι κανόνε, λαμβάνει ήδη χώρα. Ήδη υπάρχει επαρκής βαθμός ενοποίηση των αγορών χοντρική σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον Δεκέμβριο καταφέραμε να καθορίσουμε και να μας συγκρίνουν έναν οδικό χάρτη ώστε να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της, θα έχει ενοποιηθεί, θα ενοποιηθεί σε μια ενιαία αγορά ενέργειας χονδρικής έως το 2014 και συνεχίζουμε την παρακολούθηση ώστε να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα με αυτή την, ε, την πορεία. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο προωθούμε τη διαδικασία. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, αν είχαμε κάνει αυτή τη συνάντηση πριν από τρει-τέσσερι μήνε, θα ήμουν απεσιόδοξο. Πρέπει να πω ότι ο τομέα του φυσικού αερίου έχει κινηθεί πολύ τι τελευταίε εβδομάδε και μέσα στο έτος ε, διάφορα πιλωτικά έργα θα καθοριστούν όσον αφορά τον καταμερισμό και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ θετική κίνηση, σημαντική κίνηση μάλιστα μέχρι τα τέλη του έτους. Θα μπορούμε να γνωρίζουμε η πρόοδο μπορούμε να αναμένουμε ως το 2014 ρεαλιστικά. Αλλά και πάλι πιστεύω εδώ υπάρχει η δραστηριοποίηση και ήδη αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Για τον κύριο Μπαλσίτης Συμφωνώ με αυτό που λέτε για την ευκαιρία παρακολουθήσης της αγοράς και να φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Ελπίζω να μην σας έδωσα λάθος εντύπωση όταν λέω ότι υπήρξαν προβλήματα με τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ουσιαστικά η εργασία μας είναι καταπληκτική. Εντυπωσιακά καλή οι κυβερνήσεις και ο οργανισμός είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί. Ωστόσο, έχουμε καταφέρει να βρούμε έναν ικανοποιητικό τρόπο συνεργασία με το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή εργασιακή σχέση. Βασικά αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουν αυτοί προβλήματα στις χώρες τους, πρέπει να πάνε, θέλουν να πάνε σε νέε περιοχές. Δεν είχαν μεγάλη εμπειρία στην παρακολουθήση της αγορά χονδρική και τώρα απαιτείται από αυτού να παρακολουθούν εν μέρη την αγορά, να επιβάλλουν νόμους και έχουν περιορισμένους ενδεχομένου πόρους. Έτσι λοιπόν χρειάζονται, ξέρετε, και πολλοί εμπειρογνώμονες για όλα αυτά. Υπήρξαν προβλήματα μεταξύ του... Αν υπάρχουν προ... Δεν είναι ακριβώς ότι έχουμε προβλήματα μεταξύ μας, είναι ότι αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Ωστόσο υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν και να καλύψουν τα κενά πόρων που εμείς έχουμε, γιατί και αυτοί έχουν να κάνουν με μεγάλες προκλήσεις. και αυτοί και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με τους διαθέσιμους πόρους. Ελπίζω να απάντησα ε, σε όλα τα ζητήματα. Αν μπορείτε να μου δώσετε ακόμη δύο λεπτά, διότι ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν σύντομα. Ήδη ανέφερα ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία για το πρόγραμμα εργασία. Ε, θα την ξεκινήσουμε σύντομα για το πρόγραμμα εργασία για του χρόνου. Σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια προσέγγιση εδώ στι Βρυξέλλες, την πρώτη έκθεση ετήσια δραστηριοτήτων ε, του οργανισμού. Θα διατεθεί στις 15 Ιουνίου και θα αφορά το περασμένο έτος και φυσικά θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να βρείτε λεπτομέρειες σε σχέση με το τι κάναμε μέχρι σήμερα και όλα αυτά που σας περιέγραψα σήμερα. Η αποστολή στη Λιουμπιάννα για μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προγραμματιστεί από ό,τι κατάλαβα τον Αύγουστο. Φυσικά είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι στη Λιουμπιάννα και ειδικότερα στα γραφεία μας. Με μεγάλη χαρά και εγώ και οι συναδελφοί μου θα σας συναντήσουμε εκεί. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά όλους εσάς για τη συνεχή σας στήριξη προς τον οργανισμό και την εμπιστοσύνη σας. Αυτό ε, φαίνεται σε κάθε βήμα και πολλές φορές πέραν των προσδοκιών μας. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Πολύ ωραία η σημερινή ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες μας σήμερα. Thank you very much, Mr. Uh, yes, I understand you might come back here in ITRA ε, μπορεί να επανέλθετε στην Ήτρε τον Ιούλιο να μας παρουσιάσετε πρόγραμμα εργασίας ε, για το 2013. Ε, είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. 18 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση της Ήτρε και 19 Ιουνίου επίσης. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιστροφή σε όσους έχετε ταξίδι μπροστά σας.